Και να συνεχίσουμε λοιπόν με την ε, συνεδρίασή μας. Πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη, να σας πω ότι το σημείο 5, ρύθμιση ε, με την Ελβετική Συνομοσπονδία, σχετικά με την συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Αυτό το θέμα λοιπόν της ημερησίας διατάξεως έχει ε, αναβληθεί. Συμφωνείτε? Πολύ ωραία. Επομένως, να κάνουμε άλλες ανακοινώσεις. Ε, αφορά την ε, ε, αποστολή της Επιτροπής μας στην Ιταλία την επόμενη εβδομάδα, 26-28 Μαρτίου. σύμφωνα με την παρούσα σύνθεση έχουμε τρία πλήρη μέλη και έχουμε και τέσσερις αιτήσει για συνοδευτικά μέλη από τον κύριο Γιακολίνο, την κυρία Αντζελίλη, τον κύριο Καρόνα και τον κύριο Μποργέτσιο. Ε, σύμφωνα πάντως ε, με, τους, ε, με τον εσωτερικό κανονισμό μας όσον αφορά τα συνοδεύοντα μέλη, αυτά δεν μπορούν σε αριθμό να υπερβαίνουν τον αριθμό των πλήρων μελών της αποστολής. Επομένως έχουμε τρία πλήρη μέρη, αλλά μπορούν να υπάρχουν μονάχα τρία συνοδευτικά μέλη. Επομένως θα πρέπει να ληφθεί απόφαση όσον αφορά τα συνοδευτικά μέλη τα οποία θα συμμετάσχουν σε αυτήν την αντιπροσωπεία ως επικεφαλής της αποστολής και σε συζήτηση με, δύο, με τα δύο άλλα πλήρη μέλη της αποστολής, τον κύριο Έγγελ και την κυρία Γκέντσε, προτείνουμε τα ακόλουθα μέλη να συνοδεύσουν την αποστολή μας στην Ιταλία. Ο κύριος Γιακολίλο, η κυρία Αντζελίλη και ο κύριος Καρόνα. Αν συμφωνείτε, θα επικυρωθεί η απόφαση αυτή. Πολύ ωραία, σας ευχαριστώ. Όσον αφορά τώρα το γλωσσικό καθεστώς της Επιτροπής μας, πρέπει να σας πω ότι φιλανδικά, εσθονικά, μαλτέζικα και κροατικά δεν είναι διαθέσιμα σήμερα. Σας ευχαριστώ για την κατανόηση. Περνάμε επομένω στο σημείο 6 τη ημερησία διατάξεω που αφορά την έκβαση πολιτικών διαλόγων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα στον τομέα των ιστορικών υποθέσεων. Έχουμε εδώ μαζί μας το Γενικό Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων. Έχουμε επίσης ε, τον κύριο Λορέντζο Φοντάνο, ο οποίος είναι ο εισηγητής μας, ε, ε, καθώς επίσης και την κυρία Σιλβί Γκυγιόμ για το Ταμείο Εσωτερικής, για το Ταμείο Ασύλου και τέλος όσον αφορά την ε, ε, συνεργασία, αστυνομική συνεργασία και καταπολέμηση οργανωμένου εγκλήματος, τον κύριο Ιακολίνο. Επίσης έχουμε τον κύριο Στέφανο Μανσερβίζη, ο οποίος εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο οποίος ε, θα μας κάνει μια παρουσίαση της έκβασης των πολιτικών διαλόγων σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που καθορίζει τις γενικές διατάξεις όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Οι διάλογοι Ευθύ έχουν λάβει μέρη μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών ε, μελών στα πλαίσια του καθορισμού του πολιετούς προγράμματος των ε, διαλόγου των κρατών μελών. Πρόκειται για ε, διάλογο ο οποίος εστιάζεται στα γενικά αποτελέσματα τα οποία θα πρέπει να επιτευχθούν μέσω των εθνικών προγραμμάτων έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των κρατών μελών σε, διάφορες, σε διάφορα στοιχεία τα οποία καλύπτονται από τα εν λόγω ταμεία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προετοιμάσει ένα υπόμνημα ε, και, πληροφορία, και ε, πληροφορίες σχετικά ε, με την κάθε χώρα, σχετικά με το, την έκβαση των πολιτικών διαλόγων με κάθε μία χώρα μέλος αυτό το έχει δοθεί στα μέλη της Επιτροπής μας. Θα δώσουμε λοιπόν αμέσως τον λόγο στον κύριο Στέφανο Μανσερβίζη έτσι ώστε να μας κάνει μια παρουσίαση σχετικά με την έκβαση αυτών των πολιτικών ε, διαλόγων και να μας χαράξει τις γενικές γραμμές. Ε, πρέπει να σας πω ότι ε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε τις ερωταπαντήσεις μέχρι τις 10 και 20 και μετά θα συνεχίσουμε με την παρουσίαση της έκβασης των πολιτικών διαλόγων όσον αφορά το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας και μέχρι τις 10.30. Ο κύριος Μαν Σερβίζη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση την οποία μου απευθύνατε. Έχω πει επανειλημμένα ότι το θέμα είναι σημαντικό, ο πολιτικός αυτός διάλογος είναι σημαντικός και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή βεβαίως. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα εξακολουθήσει να έχει στενές επαφές και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών αλλά και με το Κοινοβούλιο ε, γενικότερα ε, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσουμε όπως είπατε και εσείς με τον πλέον πολιτικό και στρατηγικό τρόπο τα χρήματα αυτά. Ε, και βεβαίω στα πλαίσια αυτά η διαρκή συνεργασία και επαφή το Κοινοβούλιο είναι ιδιαίτερη σημασίας. Θα συζητήσουμε λοιπόν για την έκβαση των πολιτικών διαλόγων και εγώ θα παρουσιάσω ένα δελτίο αναχώρα ε, έτσι ώστε να συνοψίσω τα κεντρικότερα ε, ζητήματα. Είχαμε 32 διαλόγους που έχουν ολοκληρωθεί ε, βάσει μιας πολλαπλής ε, ε, γεωμετρίας και που σημαίνει ότι εκτός από τις χώρες μέλη έχουμε και συνδεδεμένες χώρες με τις οποίες συνομιλούμε για τα θέματα αυτά. Να κάνω πρώτα κάποιες γενικές θεωρήσεις όσον αφορά τη διαδικασία. Θα έχετε διαπιστώσει ότι εργαζόμαστε ε, με μεγάλο ορθολογισμό γιατί βεβαίως έχουμε ε, την νομική βάση και προσπαθούμε να ε, προσπαθούμε να εργαστούμε βάσει μιας υπόθεσης για το που θα είναι όσο πιο κοντά γίνεται στη νομική βάση έτσι όπως αυτή θα μπορούσε να είχε οριστεί και βεβαίω ε, προσπαθούμε να λαμβάνουμε υπόψη μα και τα διεθνή προβλήματα. Έλεγα λοιπόν ότι έχουμε ε, μεγάλη δόση λογική ε, λήψη της νομική βάσης. Το δεύτερο σημείο είναι ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εθνικά προγράμματα. Κυρίως δε, και αυτό έχει υπογραμμιστεί επανειλημμένα από το Κοινοβούλιο, όσον αφορά το ελάχιστο ποσοστό Η το συστημα συμμορφωση αυτή ε, βασίζεται σε ένα state of play, γιατί βεβαίως ε, από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Ε, και για κάθε χώρα προσπαθήσαμε να κάνουμε μία gap ανάλυσης που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και που βασίζεται σε, κάποιες, ε, σε κάποια ειδικά στοιχεία τα οποία ε, θα πρέπει να συζητήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την κάθε χώρα έτσι ώστε να υπάρξει μια κοινή βάση μέσω της οποίας θα ταυτοποιήσουμε την κατάσταση. Θα πρέπει επίσης να οργανωθεί ο διάλογος με τρόπο ώστε να δούμε που θα έπρεπε να βρίσκονται τα κράτη-μέλη, δηλαδή ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι και ποια είναι τα επιτεύγματα τα οποία θα πρέπει να προσδοκούν οι χώρε μέλη. Τρίτο σημείο σημαντικό είναι ότι από αυτή την άποψη ε, θα πρέπει να έχουμε μία διαδικασία η οποία δεν θα βασίζεται μονάχα σε διαδικαστικά στοιχεία ε, αλλά στο μέτρο του δυνατού ε, να ορίζεται από τους στόχους που θέλουμε να πάμε και ποιοι, που θέλουμε να φτάσουμε. Αυτό ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο στην ταυτοποίηση των στόχων του διαλόγου και η στόχοι του διαλόγου ήταν κυρίως να υπάρχει μια κοινή ε, κατανόηση κάποιων θεμάτων έτσι ώστε ε, κάποια στιγμή ε, να έχουμε μια κοινή ανάγνωση των στοιχείων αυτών Βεβαίως αυτή η ταύτιση απόψεων δεν επετεύχθη πάντα και δεν μπορέσαμε να έχουμε συμφωνία επί όλων των λεπτομεριών, αλλά βεβαίως να έχουμε μια ε, γενική εικόνα η οποία ε, θα οδηγείται, ε, θα έχει κεντρικό της όχημα την πολιτική και τους στόχους του, τι πρέπει να κάνει ο καθένας. Βεβαίως θα επανέλθω με λεπτομέρειες όταν θα μιλήσουμε για το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης. Ο άλλος στόχος είναι ότι πρέπει να υπάρχει ε, το θέμα, το θέμα το οποίο είναι ευαίσθητο, το θέμα της ιδιοκτησίας σε επίπεδο ε, ευρωπαϊκών ε, χωρών. Ξέρετε ότι, και δεν θα σας το πω εγώ, ξέρετε ότι το θέμα της, κτήσης, της ιδιοκτησίας συγγνώμη, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ε, λοιπόν, πώς αξιολογώ εγώ την έκβαση των πολιτικών αυτών διαλόγων. Πρώτον, ε, τις ε, αξιολογώ πάρα πολύ θετικά, γιατί ο στόχος της απλούστευσης της αρχιτεκτονικής και του συστήματος ε, έπρεπε να ταυτοποιηθεί και από τις ίδιες τις χώρες, τα κράτη-μέλη, και αυτό δεν είναι προφανές. Επομένως, αυτή η διαδικασία της απλούστευσης της συζήτησης ε, που βασίστηκε στο ακριβώς τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας έβγαλε το βάρος της γραφειοκρατίας από πάνω μας και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης ε, αντιμετωπίστηκαν ε, και κάποιες ελλείψεις εμπιστοσύνης γιατί ξέρετε ότι από την αρχή δεν ήταν όλες οι χώρες ανοιχτές σε αυτόν τον πολιτικό διάλογο γιατί πολλοί είπαν αυτή είναι η δικιά μας δουλειά. Δεν πρέπει η Κομισιόν να ανακατευτεί αλλά στο τέλος ε, ε, είναι προφανές ότι αν εμείς πρέπει να εγκρίνουμε στο τέλος της διαδικασίας το εθνικό πρόγραμμα, οπωσδήποτε θα πρέπει να συνεργαστούμε. Ε, προσπαθήσαμε λοιπόν να ξεπεράσουμε αυτήν την έλλειψη εμπιστοσύνης, προσπαθήσαμε να καλύψουμε τα κενά και τις αποστάσεις που μας χώριζαν. Και πρέπει να σας πω ότι παρά τις αρχικές δυσκολίες, στο τέλος όλα ήταν διαφανή και πολύ ωραία. Ε, η τελευταία μου γενική αξιολόγηση είναι ότι τελικά καταφέραμε να επιτύχουμε και καλές συμφωνίες όσον αφορά τους δείκτες ε, ή μάλλον όσον αφορά την αρχή ε, ε, εγκαθίδρυσης τέτοιων δικτών βάσει ενός διαρκούς πολιτικού διαλόγου μέσω του οποίου θα βλέπουμε τι δεν έχουμε επιτύχει, τι έχουμε επιτύχει και πώς μπορούμε να πάρουμε και ποια θα είναι τα διορθωτικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν. Νομίζω ότι σε γενικές γραμμές η έκβαση είναι θετική. Θα τα πούμε βέβαια και αυτά, αλλά νομίζω ότι ε, ε, η διαδικασία έχει διευκολύνει τον στόχο τον οποίο θέλουμε εν τέλει να επιτύχουμε. Είπαμε ότι είχαμε κάποιες ε, συμφωνίες όσον αφορά τις τάσεις, άλλωστε δεν χρειάζεται να με γιατί ξέρετε σας έχω δώσει και τα δελτία αναχώρα. Όσον αφορά το Ταμείο Σύλλου Μετανάστευσης, κυρίως όσον αφορά το άσυλο, είχαμε, η εικόνα είναι καθαρή. Έχουμε δύο ομάδες χωρών. Έχουμε την ομάδα χωρών οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες γιατί υφίστανται μεγάλες πιέσεις ε, και ε, τις χώρες οι οποίες λόγω της γεωγραφικής τους ε, θέσης βρίσκονται υπό φυσική πίεση ή κινδυνεύουν να έχουν μεγάλη πίεση όσον αφορά και την νόμιμη μετανάστευση και τους ετούντες άσυλο βεβαίως ε, αυτές οι χώρες θα πρέπει οπωσδήποτε να εγκαθιδρύσουν ένα σημαντικό, σωστό σύστημα έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν και τα μεγάλα νούμερα των ετούντων άσυλο αλλά και τα μεγάλα νούμερα των νομίμων μεταναστών. Επίσης έπρεπε να συμφωνήσουμε ε, σχετικά με τα όρια και τα σχέδια τα οποία ε, θα αφορούν τις ποσοστώσεις και τα όρια καθώς επίσης και οτιδήποτε απορρέει από τη συμφωνία του Δουβλίνου. Ε, και βεβαίω εκεί έχουμε δυσκολίες όσον αφορά την δυνατότητα υποδοχής, όσον αφορά ε, την ε, βοήθεια, όσον αφορά την αντιμετώπιση των νομίμων και μη νομίμων μεταναστών κτλ. Οπωσδήποτε εκεί θα πάνε πολλά από τα χρήματα τα οποία θέλουν να δαπανίσουν οι χώρες, αλλά υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των χωρών. Δεύτερο θέμα, το θέμα της ένταξης. Εδώ είχαμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση ε, όσον αφορά την ένταξη των ετούντων άσυλο, που ξέρετε ότι είναι μια ειδική κατηγορία Εκεί ε, μπορέσαμε να βρούμε κάποιες ε, ε, success stories που υπάρχουν σε διάφορες χώρες, αλλά και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε όλες τις υπόλοιπες. Και νομίζω ότι εκεί η διαφορά ήταν σαφής ανάμεσα σε την ομάδα χωρών που έχουν συνηθίσει να αντιμετωπίζουν αυτές τις μεγάλες ροές μεταναστών, παρανόμων μεταναστών και τον άσυλο και τους, την ομάδα των νέων χωρών που δεν είχαν έτσι εμπειρία πάνω στο θέμα αυτό και έπρεπε βεβαίως να ανταλλαγούν οι καλύτερες πρακτικές, τα μαθήματα, ε, τα νέα στοιχεία κτλ. Και εδώ είχαμε δύο θέματα τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Ένα, πώς, ε, ε, μπορεί να, πώς μπορούμε να εγγυηθούμε, να την πρόσβαση στην ελεύθερη αγορά και πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε την πρόσβαση των νομίμων μεταναστών σε αυτήν την αγορά. Το δεύτερο, το οποίο μου άρεσε και πάρα πολύ, ήταν ότι ε, έγιναν δύο ε, συνέργειες ε, με, τα διαφορετικά ταμεία. Γιατί, είχαμε, γιατί η συνεργασία μεταξύ του Κοινωνικού Ταμείου και του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης πρέπει να είναι μεγάλη και βεβαίως είναι ένα μικρό ταμείο σε σχέση με τα διευθυντικά ταμεία και επομένως επιτόπου είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν συνέργειες και μάλιστα με συγκεκριμένο αυτό τρόπο που άλλωστε πρέπει να πω ότι έχουν ε, ε, έχουν επιβεβαιώσει την αρχική μας άποψη σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργήσει η συνεργασία σε πρακτικό επίπεδο και επιτόπου. Το θέμα της ε, επιστροφής ε, επίσης ε, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Το να γίνει αποτελεσματική η πολιτική επαναπρόθεση είναι πάρα πολύ σημαντικό έτσι ώστε σιγά σιγά να προχωρήσουμε σε ένα καθεστώς εθελούσιας επιστροφής στις χώρες μέσω συνεργασίας κρατών μελών και διεθνών οργανισμών όπως τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης κτλ. Αλλά και με τρόπο ώστε να δημιουργηθεί μια πραγματική στρατηγική για τις ε, επιστροφές. Γιατί αν δει κανείς ε, το, τους μετανάστες ε, οι οποίοι καθορίζονται ως παράνομοι και τον αριθμό των μεταναστών που αποφασίζουν να επιστρέψουν, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο χάσμα και επομένως θα πρέπει η βοήθεια που θα δοθεί στην επιστροφή αυτή να είναι πολύ σημαντική. Τώρα το θέμα της επαναπροώθησης και αυτό είναι πολύ σημαντικό και για την Κομισιόν και για τα κράτη-μέλη. Είδαμε μια αρχική ε, καλή διάθεση έτσι ώστε όλοι να παίξουν το παιχνίδι και να δοθούν και επιπλέον χρήματα και επομένως ε, ενδεχομένως θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα ειδικά σε κάποιες ε, περιοχές και σε κάποιες εποχές οι οποίες δίνουν μεγαλύτερη πίεση. Αυτά είναι τα κεντρικά στοιχεία τα οποία μας απασχολούν όσον αφορά το Ταμείο Σύλλου Μετανάστευσης και βεβαίως ε, εξειδικευμένα θα δείτε και τα δελτία τα οποία σας έχω μοιράσει αναχώρα. Τώρα, ε, έχουμε από τη μία πλευρά το θέμα των ε, συνόρων και εδώ νομίζω ότι είναι τρεις οι στόχοι οι οποίοι είναι κοινοί για όλους έστω και αν η ποσολογία είναι, η δοσολογία είναι διαφορετική. Πρώτον η χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών. Αυτό νομίζω το ανέφεραν όλες οι χώρες μέλη και αυτό οπωσδήποτε θα το στηρίξουμε και βεβαίως όλοι ε, πρέπει οπωσδήποτε να διασφαλίσουμε ότι ό,τι γίνεται σε εθνικό επίπεδο θα είναι συμβατό με την ε, έκβαση της ε, ε, νομικής διαδικασίας όσον αφορά όσον αφορά τα ευφυή σύνορα. Αλλά αυτό είναι το κεντρικό εργαλείο το οποίο θα, στο οποίο θα πρέπει να επενδύσουν όλοι. Δεύτερον, όσον αφορά το, την διαχείριση των σύνορων και αυτό είναι ε, σημαντικό γιατί τον ρόλο που θα παίξει ο Νοσούρ για, το, τη διαδικασία ε, είναι, και αυτό, είναι και αυτό σημαντικός και θα είναι ε, σημαντικό το πώς θα επενδύσουν τις ικανότητες τους, την τεχνολογία τους οι χώρες μέλη και πώς θα συνεργαστούν με όρους εμπιστοσύνης. Και επίσης τρίτο σημείο η προξενική συνεργασία τι, ε, με ποιο τρόπο θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε ε, να αντιμετωπίσουμε το σύστημα ε, των θεωρήσεων Σέγγεν. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το θέμα έτσι ώστε οι διαδικασίες ε, για τις ε, θεωρήσεις, ε, για τη βίζα να είναι κοινέ. Και βεβαίως προβλέπονται και μια σειρά διαδικασιών οι οποίες θα βελτιώσουν την κατάσταση, θα απλουστεύσουν την κατάσταση και θα βελτιώσουν την κατανόηση. Όσον αφορά τώρα το Ταμείο για την Εσωτερική Ασφάλεια και την Αστυνομία, νομίζω ότι το κυριότερο θέμα ήταν ότι ήταν η πρώτη φορά πραγματικά που ζητήθηκε από τα κράτη-μέλη ε, να καθορίσουν πολιετή στρατηγική για την ασφάλεια. Γιατί μέχρι τώρα, όπως καλά γνωρίζετε, ε, μόνο με μονομένα προγράμματα στήριζαν το θέμα αυτό και επομένως η έλλειψη εμπιστοσύνης αλλά και η ε, φυσική τάση βάση δυσπιστίας ε, και δισταγμού που έχουν τα κράτη-μέλη να ανοιχτούν σε θέματα εσωτερικής ε, ασφάλειας. Αυτά ήταν τα δύο κεντρικά σημεία δυσκολίες και δεν σας κρύβω ότι ε, έπρεπε να καταβληθούν πιο συγκεκριμένες προσπάθειες και να καταβληθούν και στο μέλλον βεβαίως. Οπωσδήποτε τα κράτη-μέλη πρέπει να προετοιμάσουν πολιετές πρόγραμμα ασφάλειας ε, και σε αυτό συμφώνησαν όλοι και νομίζω ότι βρήκαμε και τον τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα πρώτον ε, ταυτοποιώντας τις ε, προτεραιότητες και δεύτερον επιμένοντας στην συμπληρωματικότητα. Και φαίνεται ότι αυτό είναι δυνατόν να γίνει ε, με, τον, την ταυτοποίηση με τον στόχο που βασίζεται στην ανάλυση της όχτα που έχει κάνει η Europol. Και γύρω από αυτά, τα βασικά θέματα που επισημάνθηκαν στο διάλογο ήταν να ασχοληθούμε με το χαμηλό επίπεδο κατάρτισης των αρχών επιβολής του νόμου το οποίο ήταν αναμενόμενο. Όλα τα κράτη-μέλη ήθελαν να επενδύσουν σε αυτήν την δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι θα πρέπει να έχουμε κάποια ευελιξία όσον αφορά την κατάρτιση. Έχουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο κομμάτι της ε, κατάρτισης. Κατόπιν έχουμε την ε, διασυνορική καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Ο βασικός άξονας όπου υπήρχε σύγκληση ήταν να αντιμετωπίσουμε την καταπολέμηση των ναρκωτικών, ιδιαίτερα των νέων ναρκωτικών, ε, αυτών που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι συνθετικά κτλ, αλλά και να βελτιώσουμε τη συνεργασία, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Δεύτερον, η καταπολέμηση του κυβερνοεγκλήματος. Αυτό είναι νέο στοιχείο, είναι μια αναδυόμενη πτυχή του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας. Γι' αυτό το κυβερνοέγκλημα και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν άλλον έναν τομέα στον οποίο πιστεύουμε ότι θα προσανατολίσουν τα κράτη-μέλη τα προγράμματά τους και τρίτον ε, το εμπόριο ανθρώπων. Η ε, εμπορία ανθρώπων και όλα αυτά συνδέονται μεταξύ τους η εμπορία ανθρώπων, το εμπόριο ναρκωτικών ε, και το λαθρεμπόριο όπλων. Είναι λοιπόν και αυτό ένα τρίτο ε, πρόβλημα το οποίο είδαμε. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να κλείσουμε με κάθε κράτος μέλος ε, τον κύκλο αυτό, διότι τι επίκειται. Θα πρέπει να υποβληθεί το εθνικό πρόγραμμα και μέχρι στιγμής θα ήθελα να τονίσω δεν έχουμε λάβει κανένα διότι δεν ισχύει ο κανονισμός, διότι χρειάζεται χρόνος να αφομοιώσουν τα στοιχεία αυτά, διότι όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια, Συχνά πρέπει οι κατακαιρματισμένες διοικήσεις να υποβάλουν συντονισμένη θέση. Γι' αυτό λοιπόν συνεχίζουμε να ασκούμε πίεση όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά η προσδοκία μας είναι να έχουμε τα προγράμματα αυτά μέχρι τον Ιούλιο ή να ξεκινήσουμε να λαμβάνουμε τον Ιούλιο που θα έχει τεθεί σε ισχύ η νομική βάση και που θα μπορέσουμε να εξετάσουμε τα προγράμματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε λάβει τίποτα επί της ουσίας, αλλά δεν έχουμε λάβει επίσημο εθνικό πρόγραμμα. Γίνεται όμως ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα συστατικά στοιχεία των εθνικών σχεδίων. Και γι' αυτό η πρόβλεψή μας είναι Εάν συνοχιστούν έτσι οι εργασίες θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε να εγκρίνουμε τα προγράμματα το τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς για να τα έχουμε ολοκληρώσει όλα την 1η ε, Ιανουαρίου του 2000, ε, ε, συγγνώμη, στο πρώτο εξάμεινο του 2015. Αξίζει τον κόπο να κάνουμε αυτή τη δουλειά, διότι αυτό που θέλαμε από την αρχή, να μιλήσουμε επί της ουσίες και να έχουμε κάτι που να βασίζεται περισσότερο στην πολιτική παρά στις ε, διαδικασίε είναι πολύ σημαντικό. Α συνεχίσουμε λοιπόν τη συνεργασία μεταξύ μα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο να συνεχίσουμε τον διάλογο αυτό. Τον διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με εσά δηλαδή. Για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα αποτελέσματα αυτής της διαδικασίας. Θα κλείσω εδώ και είμαι στη διαθεσή σας να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ε, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε τώρα λίγη ώρα για συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό αφού ακούσαμε την παρουσίαση του κυρίου Μασεβίση και κατόπιν θα προχωρήσουμε στο δεύτερο μέρος, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχουν κάποιοι ευρωβουλευτές που έχουν κάποιες παρατηρήσεις. Η κυρία Γκίγιομ, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και σας ευχαριστώ για την παρουσίαση αυτή, ε, η οποία γίνεται ενώπιον ε, μικρού αριθμού βουλευτών και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Ε, ευχαριστούμε για την παρουσίασή σας. Ε, τον τελευταίο μήνα είχαμε, ή μάλλον τους τελευταίους μήνες είχαμε πολύ ε, πυκνή συνεργασία και νομίζω ότι σωστά συνοψίσατε τα διακυβέρματα του διαλόγου όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα, άρα δεν θα επανέλθω από αυτόν. Έχω όμως κάποια ερωτήματα να σας υποβάλω ε, και γενικά και ειδικά όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης. Ε, για το αν κατάλαβα καλά δεν έχετε ακόμα λάβει κανένα εθνικό πρόγραμμα πλευρά κρατών μελών. Αυτή είναι μια ερώτηση. Μου το επιβεβαιώνετε συγκατανεύοντας, για τις κεφαλής. Άρα το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι συζητήσαμε πολύ ε, για τα ελάχιστα ποσοστά και νομίζω ότι στην διάρκεια του διαλόγου και πριν την ολοκλήρωσή του θα πρέπει οπωσδήποτε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά τα ελάχιστα ποσοστά θα γίνονται σεβαστά από τις χώρες μέλη, γιατί αυτό ε, το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό. Εάν αυτό δεν επιτευχθεί, θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν πληροφορίες σχετικά με την αιτιολόγηση αυτής, αυτού του μη σεβασμού των ελαχίστων των ποσοστών. Εάν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τοποθετηθεί θετικά όσον αφορά ε, αυτόν τον μη σεβασμό των ελάχιστων ποσοστών θα πρέπει να αιτιολογήσει τη θέση της. Ξέρετε καλά ε, τι εννοώ, γιατί έχουμε συζητήσει επανειλημμένα πάνω σε αυτό, δεν επανέρχομαι. Το δεύτερο στοιχείο, το οποίο θα πρέπει με προσοχή να αντιμετωπίσουμε, είναι το θέμα της διαβούλευσης ε, με τους διαφορούς διεθνεί οργανισμούς, μη κυβερνητικέ οργανώσεις κλπ. Και αυτό μας είναι ιδιαίτερα προσφυλές, όπως ξέρετε. Έχετε σε αυτή τη φάση κάποια επιστροφή όσον αφορά το διάλογο που είχατε με τα κράτη-μέλη, πώς το βλέπουν τα κράτη-μέλη και βεβαίως εάν είχατε και ε, επαφή με τέτοιους οργανισμούς, ποια είναι η δικιά τους άποψη. Και μια γενική παρατήρηση ακόμα. Εάν δεν κάνω λάθος, δεν άκουσα πολλά όσον αφορά τις ε, ε, διαδικασίες οι οποίες χρηματοδοτούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ ε, δεν τα συζητήσατε αυτά. Αν ναι, μπορείτε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες όσον αφορά αυτό το σκέλος. Ε, το Ταμείο για την Μετανάστευση αναφερθήκατε ε, σε ομάδες ε, κρατών τις οποίες χωρίσατε ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης του συστήματος ασύλου που έχουν. Ωστόσο, καλό θα ήταν να μας πείτε ποιες είναι αυτές οι χώρες, ονομαστικά δηλαδή, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες αποτελούν την, τις διάφορες ομάδες στη δεύτερη ομάδα, είπατε, αναφερθήκατε σε μια δεύτερη ομάδα, η οποία έχει συστήματα ασύλου αρκετά αναπτυγμένα, έστω και αν δεν μπορούν αυτά τα συστήματα να αντιμετωπίσουν ε, τις ε, ε, ροές των ετούντων. Και εδώ διαβάζω ε, ότι πρόκειται για χώρες ε, οι οποίες ε, δεν είναι πολύ ελκυστικές είτε γιατί δεν έχουν ικανό αριθμό μεταναστών της ίδιας κοινότητας είτε γιατί δεν έχουν ελκυστικό σύστημα κοινωνικών ευεργετημάτων. Αυτό, αυτή η διασύνδεση που κάνετε ανάμεσα στους ετούντες άσυλο που κατά κάποιο τρόπο θα κάνουν ένα social benefit shopping που θα προσπαθούν να βρουν την χώρα με το καλύτερο κοινωνικό σύστημα με προβληματίζει αυτή η ορολογία που χρησιμοποιείτε. Λίγο με προβληματίζει αν μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό. Επίσης, όσον αφορά τις επιστροφές, πάντα για το Ταμείο Σύλλου Μεταναστεύσης, ε, όσον αφορά την εθελούσια επιστροφή βρίσκω ιδιαίτερα ε, θετική αυτή την, αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης της Κομισιόν όσον αφορά τις επιστροφές ε, και όσον αφορά την πυθό την οποία επιτύχατε. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια. Είναι ενδιαφέρον να δούμε σε τι αντιδρούν θετικά οι χώρες και σε τι όχι. Επίσης, όσον αφορά τη χρηματοδότηση στις συζητήσεις μας ε, είχαμε ε, αναφέρει τις δυσκολίες πρόσβασης ε, χρηματοδότησης κυρίως για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τον τρόπο χρηματοδότησης. Τουλάχιστον αυτό είδαμε στην προηγούμενη χρηματοδοτική περίοδο και τον τρόπο με τον οποίο ολοκληρώθηκε αυτή η περίοδος. Επίσης είπατε ότι οι χρηματοδοτήσεις θα ήταν διαθέσιμες ήδη, ωστόσο ε, από ό,τι μαθαίνω οι ενδιαφερόμενοι ε, εκφράζουν μεγάλη ανησυχία, στη Γαλλία τουλάχιστον γιατί με αυτούς έρχομαι σε επαφή, ε, φαίνεται ότι πριν από το τρίτο τρίμηνο του 2014 δεν θα έχουν χρηματοδότηση όσον αφορά όμως ε, δαπάνες τις οποίες ήδη θα έχουν ολοκληρώσει μέχρι το 2014. Φαίνεται ότι δεν προτείνεται κάποια, πρόταση, δεν γίνεται κάποια πρόταση όσον αφορά ε, την ενδιάμεση περίοδο. Επομένως, ε, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία στους ε, οργανισμούς, στους διάφορους, διάφορες οργανώσεις, οι οποίες δεν έχουν την χρηματοδοτική ικανότητα να καλύψουν αυτή την ενδιάμεση περίοδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θα δαπανούμε για να ελέγξουμε κατά πόσον ε, είναι αληθή αυτά που ισχυρίζονται οι αιτούντες άσυλο ή απλώς δεχόμαστε αυτό που μας λένε ότι δηλαδή κινδυνεύουν στη χώρα προέλευσής τους. Αρκεί απλά και μόνο να καταδείξουν ότι η χώρα τους είναι επικίνδυνη ή πρέπει να αποδείξουν ότι αυτοί θα κινδύνευαν ιδιαίτερα λόγω της θρησκείας τους, της ε, εθνότητάς τους, της γλώσσας τους ή οτιδήποτε. Αναφερθήκατε ότι στην χρηματοδότηση που δίνεται για την επιστροφή αυτών που θα μπορούσαν να θεωρηθούν ε, λάθρομετανάστες ή ενώσεις τους αποκαλείται παράτυπους μετανάστες ή αυτή των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί. Πόσα προϋπολογίζονται και πόσα θα πανώνται για αυτή την επιστροφή και πέρα από τα πόσα. Ποια είναι η διαδικασία επιστροφής, τους δίνουμε απλώς εισιτήρια ή την τιμή του εισιτηρίου ή απλώς τους παρακαλούμε να φύγουν όπως ε, μας είπε πριν από δύο χρόνια ένας εκπρόσωπος της Frontex χωρίς να γίνεται κανένας έλεγχος για το εάν όντως αποχωρούν και επιστρέφουν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ζίπελ. Ευχαριστώ. Να αναφερθώ σε εντελώς άλλα θέματα. Κύριε Μαντσέρβιζη, αναφερθήκατε στα ευφυή e e σύνορα και πρέπει να πω ότι δεν είμαι απλώ εκνευρισμένη, είμαι έξαλλη. Η Επιτροπή μα έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφέ ότι είμαστε ιδιαίτερα επικριτικοί έναντι αυτού του συστήματο και αυτό ισχύει για όλες τι ομάδες ε, με πολλά διαφορετικά επιχειρήματα γιατί δεν ε, είμαστε πεισμένοι ότι έχει έννοια. Παρ' όλα αυτά η Κομισιόν το αναφέρει πάντα και πάντα ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν αυτό το σύστημα. Άρα νομίζω ότι δεν ενδιαφέρεται καθόλου η Κομισιόν για την άποψή μας, θέλει να δημιουργήσετε τελεσμένα, έστω και αν εμείς είμαστε εντελώς και κατηγορηματικά και όλοι εναντίον. Γιατί έτσι δημιουργεί καταστάσεις με τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ μετά από αυτό που είπε η Μπίρκιτ, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που έρχεται να μας ενημερώσει η Κομισιόν για την εφαρμογή και χρήση των πιστώσεων για τα ταμεία και χαιρόμεθα που έχουμε λάβει τα έγγραφα από πριν, ότι μπορέσαμε να τα δούμε. Μια λοιπόν πολύ απλή, ίσως απλοϊκή ερώτηση. Παρ' όλα αυτά έχει σοβαρή πολιτική διάσταση. καταλαβαίνουμε καλύτερα πώς δαπανούμε αναστόχο της πιστός των ταμείων. Θα μπορούσατε να μας δώσετε ποσοστά για κάθε προτεραιότητα στα διάφορα κράτη-μέλη δαπάνησης ε, των κονδυλίων. Για παράδειγμα, ή μάλλον να πω καλύτερα, τι ποσοστό των πόρων των ταμείων δίνονται για την ένταξη, για το άσυλο, για την επιστροφή, ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μην δαπανούν όλα τους τα κονδύλια για μία μόνο προτεραιότητα. Να υπάρχει μία καλύτερη κατανομή. Χαίρομαι για αυτή την παρουσίαση, αλλά λυπάμαι για το ότι αν και εμείς επιμείναμε ιδιαίτερα να έρθει η Κομισιόν να μας κάνει μια παρουσίαση και αποτίμηση, από όλα αυτά διαπιστώνουμε ότι οι παρόντες είναι τρει και ο κούκο. Ενώ είχαμε επιμείνει τόσο πολύ να έρθετε να μα τα πείτε. Συμφωνώ λοιπόν και εγώ ότι θα έπρεπε στο μέλλον να υπάρχουν περισσότεροι για να μπορέσουμε και στο μέλλον, πέρα από τη σημερινή συνάντηση, να ξεκολουθήσουμε να παρακολουθούμε τη χρήση των πόρων, ανά ποσοστό και ανά από τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ πολύ. Δεν βλέπω άλλους. Όχι. Ο κύριος Μανσερβίση για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Λέει ο κύριος Μανσερβίζη. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις που θα μπορούσα να συνδυάσω απαντώντας. Για παράδειγμα, η ερώτηση της κυρίας Γκυγιόμ και εντελώς τελευταία ερώτηση για τα ποσοστά. Έχουμε προτείνει ποσοστά και έχουμε πει ότι αν δεν γίνουν σεβαστά θα ζητήσουμε εξηγήσει. Αλλά δεν λάβαμε από πλευρά κρατών μελών προτάσεις για τα ποσοστά, για το πώς προτίθενται να κατανείμουν τις πιστώσεις. Μετά το διάλογο δεν λάβαμε ένα πίνακα που να λέει ορίστε 20% θα δώσουμε για το άσυλο κτλ. Γιατί ο διάλογος, ξέρετε, ήταν πρώτα απ' όλα για να υπάρξει περισσότερη αλληλοκατανόηση. Άρα δεν μπορώ τώρα να σας δώσω ποσοστά, γιατί κανένα κράτο μέλος δεν ανέλαβε σαφείς δεσμεύσει. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή σας και το Κοινοβούλιο να συνεχίσουν να... Ε, αυτόν τον διάλογο μαζί μας, γιατί όσο θα ε, εξετάσουμε πιο λεπτομεριακά τα προγράμματα των κρατών μελών, τόσο περισσότερο θα καταλάβουμε. Γιατί ο κανονισμός προβλέπει ποσοστά τα οποία πρέπει να, να τηρηθούν και θα πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί αν δεν τα τηρήσουν. Τότε θα είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι. Σε αυτό το στάδιο τώρα είπα, επιχειρήσαμε να μας δώσουν στοιχεία για τα ποσοστά, αλλά σχεδόν κανείς δεν μας έδωσε. Δεν μας απάντησαν συγκεκριμένα. Υπήρξαν κάποιες ακραίες περιπτώσεις. Να αναφερθώ σε παραδείγματα. Στο διάλογο, για παράδειγμα, με την Ολλανδία, οι αρχές της χώρας μας είπαν δεν θα χρησιμοποιήσουμε κανένα Ευρωπαϊκό Ταμείο για τις ε, προσπάθειες ένταξης. Και εμείς τους είπαμε ότι θα ελέγξουμε τι κάνετε, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιήσετε τους πόρους. Όχι όσον αφορά τι εθνικές επιλογές για την ένταξη, γιατί ξέρετε ότι δεν έχουμε αρμοδιότητες ε, για τα θέματα αυτά, θα ήταν παράλογο. Αλλά για να υπάρχει μια συνέπεια. Η συζήτηση λοιπόν ήταν απλώς ε, αμοιβαία ενημερωτική. Θα δούμε βέβαια τι θα περιλαμβάνουν τα προγράμματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο σε αυτό το στάδιο. Κάτι άλλο τι είδος διαβούλευση κάναμε με την κοινωνία των πολιτών, όχι μόνο με αρχές κυβερνητικές, αλλά με μη κυβερνητικούς οργανισμούς και άλλους. Κάθε φορά που είχαμε διάλογο για την πολιτική στον τομέα αυτό, προσπαθήσαμε πριν, κατά και μετά, να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών της χώρας αυτής. Και κάναμε αρκετές συζητήσεις και εδώ στις Βρυξέλλες. Με διάφορα κινήματα, πλατφόρμες, μέσω των οποίων εκπροσωπείται η κοινωνία των πολιτών. Θα δούμε το αποτέλεσμα βέβαια. Όσον αφορά τη διάθεση κονδυλίων υπάρχει πρόβλημα. Διότι οι μικρές οργανώσεις πολύ συχνά εξαρτώνται από την ε, συνέχιση της χρηματοδότησής τους. Και όταν αποφασίσαμε για τις προοπτικές ε, δημιουργείται μια διαφορά φάσης. Είπαμε επίσης ότι δεν έχουν ακόμη ε, δημιουργηθεί οι νομικές βάσεις και οι δημοσιονομικοί κανόνες σημαίνουν ότι μπορεί μέχρι το 2016 να μην μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε κάποιες οργανώσεις. Δεν μπορούμε εμείς να επεχρώσουμε τα κρατη να δώσουν προκαταβολές. Αυτό που θα κάνουμε οπωσδήποτε είναι ότι κάποιες πιστώσεις που διαχειρίζεται απευθείας η Κομισιόν και όπου προετοιμάζουμε τώρα το πολιετές μας πρόγραμμα και το πρόγραμμα εργασιών για το 2014-2015 εκεί υπάρχει και ένα τμήμα για την κοινωνία των πολιτών που θα αξιοποιήσουμε για πόρους βεβαίως που ε, διαχειριζόμεθα εμείς ε, κεντρικά για να επιτρέψουμε μέσω συγχρηματοδοτήσεων να κάνουμε ό,τι μπορούμε, ε, να εκμεταλλευτούμε όσο μπορούμε την αύξηση του του ορίου συγχρηματοδότηση που έχει περάσει το 75% όπως Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδυάσουμε τα διάφορα μέσα στη διάθεσή μας. Τώρα, ποιες είναι αυτές οι ομάδες χωρών και η ορολογία που χρησιμοποιώ. Ίσως η ορολογία μου να μην είναι η πολιτικά ορθή πάντα. Αλλά προσπαθώ ε, να περιγράψω όσο ε, ακριβέστερα γίνεται την πραγματικότητα, την πραγματικότητα αυτών που ετούνται άσυλο. Και έχω την ε, εντύπωση ότι έχουν αυτή την τάση να κάνουν αυτό το shopping, να διαλέγουν δηλαδή. Ξέρουν πολύ καλά σε ποια χώρα τι δίκαιο επικρατεί και σε ποια χώρα τι επιδόματα υπάρχουν. Για παράδειγμα, η Γερμανία και η Σουηδία διαπιστώνουν ε, ότι υπάρχουν πολλές αιτήσει ασύλου και υπάρχει τάση και αυτών που μπαίνουν από άλλη χώρα να πάνε σε αυτές τις χώρες. Ακόμη και από τα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν λέμε ότι εμείς συμφωνούμε με αυτή την πραγματικότητα, αλλά είναι η πραγματικότητα. Και εγώ πάντα αρνήθηκα να παίξω το παιχνίδι να πούμε ότι κοιτάξτε, ε, μειώστε τα επιδόματα που δίνετε για να μειώσετε την ελκυστικότητά σα. Πρώτα απ' όλα δεν έχουμε αρμοδιότητα για να το κάνουμε, αλλά νομίζω ότι δεν είναι και αξιοπρεπέ αυτό. Νομίζω ότι οι άλλες χώρες θα έπρεπε να αυξήσουν τις κοινωνικές του παροχέ. ούτω ώστε οι ετούντες άσυλο να ε, έχουν καλύτερη τύχη γιατί είναι προς το όφελος των χωρών γιατί οι λαμβάνοντες άσυλο είναι μια κοινωνική επένδυση. Πρέπει να χρησιμοποιούμε ορολογία που να είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Βέβαια δεν θέλουμε να κάνουμε διακρίσεις και δεν καταγγέλουμε ορισμένους, δεν κρίνουμε. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Ποιες είναι οι χώρες που υφίστανται πίεση. Είναι οι χώρες της πρώτης γραμμής. Στη Μεσόγειο. Η Ιταλία, η Κύπρος, η Βουλγαρία τώρα, ξέρετε πολύ καλά η Ελλάδα βεβαίως, ανέκαθεν. Αλλά προσπαθούμε να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και βελτιώνεται η κατάσταση. Οι χώρες αυτές, όπως και το Λουξεμβούργο, διαπιστώνουν μεγάλη αύξηση των ετούντων άσυλο που έχουν πολύ μικρή πιθανότητα βέβαια να γίνουν ε, δεκτές οι αιτήσει. Και στη Γαλλία εφίσταται πίεση το σύστημα και υπάρχει ε, προσπάθεια μεταρρύθμισης του για να έχει καλύτερη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Υπάρχουν χώρες που παρά την πίεση που υφίστανται τα κατάφεραν να, το, να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις. Για παράδειγμα η Αυστρία, η Ολλανδία λειτουργεί το σύστημα. Και στη Γερμανία λειτουργεί το σύστημα. Και στη Σουηδία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να κάνουν τίποτα. Αντίθετα, είναι λόγος ούτως, είναι λόγος για με βάση την πείρα αυτών των χωρών λόγω της εσωτερικής κινητικότητας να προετοιμάσουμε την εφαρμογή του άρθρου 33. Βεβαίως όλοι πρέπει να έχουμε σχέδια για έκτακτες ανάγκες. Δεν κατάλαβαν όλη την ανάγκη να τα εκπονήσουν ταχύτατα, αλλά τέλος όλοι το κατάλαβαν. Δηλαδή, το γεγονός ότι μια χώρα από τις 28 δεν είναι προετοιμασμένη μπορεί να θίξει όλες τις άλλες. Και έχουν συμβεί αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των δύο ομάδων κρατών. Αλλά ε, σε κάθε χώρα υπάρχει διαφορετικό επίπεδο επένδυσης, αντιμετώπισης. Αλλά να δούμε τώρα. Θα δούμε όταν θα δούμε τα σχέδια προγραμμάτων που θα μας υποβάλουν. Τώρα για τις επιστροφές. Δεν έχουμε κανένα μαγικό μέτρο. Αλλά τι κάνουμε. Με αποφασιστικότητα και καταλαβαίνοντας και το μήνυμα που μας αποστήλατε ως Κοινοβούλιο, προωθήσαμε στο μέγιστο την εθελουσία επιστροφή. Διό... Ξέρετε ότι και η αναγκαστική επιτροπή, επιστροφή συγγνώμη, είναι ε, απόλυτα νόμιμη και δεν είπαμε ποτέ ότι δεν θα σας στηρίξουμε αν προχωρήσετε σε ε, αναγκαστική επιστροφή που πρέπει βέβαια να σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις διαδικασίες κτλ. Αλλά η πείρα που έχουμε από την εθελουσία επιστροφή μας πείθει ότι πρέπει να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη που ε, τις επιχειρούν μέσω συνοδευτικών μέτρων. Είτε ένα ποσό χρημάτων, είτε επενδύσεις στις χώρες ε, προέλευσης και επιστροφής είναι τμήμα της εξωτερικής δαπάνης που συζητήσαμε και θα επανέλθω σε αυτό. Αυτή λοιπόν η μέθοδος είναι μια μέθοδος που θα θέλαμε να αξιοποιείται περισσότερο γιατί είναι πιο αποτελεσματική και πιο μόνιμη. Και προσπαθούμε να γίνει πιο συστηματική η χρήση αυτής της ε, εθελουσίας ε, επιστροφής. Τώρα, οι εξωτερικές ε, δαπάνες ορισμένα κράτη-μέλη είπαν ότι ένα τμήμα των ε, εθνικών χρηματοδοτήσεων, η Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, ένα τμήμα λοιπόν των ε, εθνικών χρηματοδοτήσεων για εξωτερικές δράσεις. Βεβαίως ε, το επιτρέπει η νομική βάση, είναι δυνατό. Είπαμε ότι θα πρέπει να αποφευχθεί μέσω αυτής της δυνατότητας μεγαλύτερος κατακαιρματισμός της δράσης της Ένωσης έναντι τρίτων χωρών. Και θελήσαμε να εργαστούμε μέσω εταιρικών σχέσεων για την κινητικότητα. Για παράδειγμα, οι χώρε τη Βόρεια Αφρική, Μαρόκο, την Ισία και η Λιβύη, αλλά η Λιβύη είναι σε διαφορετική κατάσταση. Οι χώρε λοιπόν αυτέ με τι οποίε έχουμε μια κοινή πλατφόρμα θα πρέπει να αξιοποιήσουν αυτή την πλατφόρμα, ώστε κάθε κράτο μέλο να πει τι θέλει να κάνει, αλλά ο καθένα, το κάθε κράτο μέλο να συνεργάζεται με τους άλλους. Να υπάρχει περισσότερη λοιπόν ε, προσπάθεια συντονισμού, ούτως ώστε και οι πόροι που κεντρικά διαχειρίζεται η Κομισιόν, που είναι το πραγματικό μέσο για εξωτερική δράση και οι πόροι που ε, διαθέτουν ε, οι γενικές διευθύνσεις που είναι υπεύθυνες για εξωτερική δράση, θα πρέπει λοιπόν, επειδή είναι περιορισμένοι οι πόροι μα, όλοι αυτοί να αξιοποιηθούν συντονισμένα, ούτω ώστε να επενδύσουμε για τη μετανάστευση και την κινητικότητα στα πλαίσια τη εξωτερική δράση Και στη Μεσόγειο έχουμε ήδη κάποια αποτελέσματα, γιατί το τμήμα μετανάστευση και κινητικότητα είναι υψηλότερο ποσοστό στα εθνικά και περιφερειακά προγράμματα της Γενικής Διεύθυνσης ΔΕΦΚΟ και των ε, συναδέλφων μας που χειρίζονται τους πόρους για την ανάπτυξη. Ελπίζουμε αυτά τα στοιχεία να συμπεριληφθούν στα προγράμματα. Όσον αφορά το ερώτημα για το πώς να διαχειριστούμε τις επιστροφές και την αρχή της ασφαλούς χώρας προέλευσης. Εάν θέλουμε να το συζητήσουμε, αυτό είναι ένα πράγμα, αλλά τώρα νομίζω μιλάμε για τον πολιτικό διάλογο, είναι διαφορετικό θέμα. Όπως και να έχει, αν θέλει η Επιτροπή σας, μπορώ να σας παρουσιάσω τις ε, δαπάνες του Ταμείου Επιστροφών μέχρι στιγμής. Αυτά έχουμε στα χέρια μας, το τι θα έχουμε στο μέλλον δεν το γνωρίζουμε, διότι δεν έχουμε λάβει ακόμα κανένα εθνικό πρόγραμμα. Είναι αδύνατον λοιπόν να πούμε κάτι για το μέλλον. Εάν όμως θέλετε τα στοιχεία αυτά κύριε Πρόεδρε, ευχαρίστω να σας υποβάλω τα στοιχεία αυτά για να γνωρίζετε τι έχει γίνει μέχρι τώρα και πώς έχουν δαπανηθεί οι πόροι. και στο βαθμό που είναι δυνατόν θα σας δώσω τα καλύτερα παραδείγματα ε, του πώς μπορέσαμε να συνοδεύσουμε τις επιστροφές αυτές με τους πόρους που έχουμε για την ε, ε, επανεγκατάσταση. Αλλά αυτή είναι άλλη συζήτηση όσον αφορά τα ευφυή e σύνορα. Γνωρίζω ότι γίνονται πολλές επικρίσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι απολύτω θεμητό, αλλά δεν μπορείτε να περιμένετε η Επιτροπή να υποβάλει μια πρόταση που να σταματάει οποιαδήποτε δραστηριότητα στο θέμα αυτό. Αν το Κοινοβούλιο αποφασίσει να μην προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό, έχει καλώ, αλλά εμεί υποβάλλουμε μια πρόταση και λαμβάνουμε όλα τα συνοδευτικά μέτρα. Το πραγματικό επίκεντρο δεν είναι εδώ, είναι στο πώς τα κράτη-μέλη μπορούν να επενδύσουν σε κάτι που να μην αντίκειται τελικά στο πιθανό αποτέλεσμα των ευφυών συνόρων. Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τα κράτη-μέλη να κάνουν αυτό που κάνουν. Το πραγματικό πρόβλημα είναι αυτό που κάνουν ήδη τα κράτη-μέλη. Διότι, αν πάμε 10 χρόνια πίσω, όταν ξεκίνησε αυτή η ιδέα των ευφυών συνόρων, οι τεχνολογίες ε, αυτές ε, στα σύνορα ήταν προνόμιο λίγων αεροδρομίων στα κράτη-μέλη, ενώ τώρα είναι κάτι που έχουν ε, σχεδόν όλα τα διεθνή αεροδρόμια στα κράτη-μέλη και σε, κάποια, και σε κάποιους συνοριακούς σταθμούς στη θάλασσα και στη στεριά. Ε, θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε τα κράτη-μέλη να τα κάνουν αυτά όλα μόνα τους χωρίς ε, κανένα βαθμό διαλειτουργικότητας ε, και χωρίς να σέβονται τον ιδιωτικό βίο σύμφωνα με τους δικούς μας κανόνες. Γι' αυτό η δική μου προσέγγιση είναι κάπως διαφορετική. Είναι ότι όσο μπαίνουμε στο παιχνίδι, τόσο μπορούμε να προσανατολιστούμε προς τους ευρωπαϊκούς στόχους. Ε, είτε με τους πόρους των κρατών μελών, είτε με δικούς μας πόρους, ε, είτε με συγχρηματοδότηση. Αλλά η νομική βάση προβλέπει ε, τις δραστηριότητες αυτές. Εάν τελικά δεν απογειωθεί το πρόγραμμα αυτό, εάν τελικά δεν λειτουργήσει, τότε ε, ας είναι, αλλά εμείς τουλάχιστον έχουμε υποβάλει μια πρόταση και ας είμαστε τουλάχιστον συνεπείς με αυτήν. Αλλά παρακαλώ να συνεχιστούν οι συζητήσεις πάνω στο θέμα αυτό για να δούμε τι θα συμπεριλάβουν τα κράτη-μέλη στα εθνικά τους προγράμματα. Άλλωστε, όπως είπα, είμαστε στην αρχή του διαλόγου αυτού, όχι στο τέλος. Και θα ξανάρθουμε και θα σας παρουσιάσουμε περισσότερα στοιχεία για το πρόγραμμα αυτό γιατί θα γνωρίζουμε και περισσότερα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ε, αναλυτικές αυτές εξηγήσεις. Νομίζω ότι καλύψαμε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Θα ήθελα να ρωτήσω τους ε, βουλευτές εάν υπάρχουν άλλες ε, παρατηρήσεις ή ερωτήσεις. Ο κύριος Μανσερβίση ε, εξέφερε τη διάθεσή του να μας υποβάλει στοιχεία σχετικά με το Ταμείο. Η κυρία Ζίπελ θέλει να κάνει μια παρατήρηση. Μία σύντομη παρατήρηση. Σημειώνω ότι η Κομισιόν θεωρεί ότι έχει δικαίωμα να εφαρμόζει προτάσεις ακόμα και όταν δεν υπάρχει σχετική απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Όχι. Ο καθένας διαδραματίζει το δικό του ρόλο σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο. Σέβομαι απολύτω τι επικρίσει, μπορεί τελικά να υπερισχύσουν, αλλά θα πρέπει και εσεί ε, να σεβαστείτε το γεγονό ότι υπάρχει μια νομική βάση σχετικά με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών στα σύνορα. Θέλουμε να αποφύγουμε τις αντιφάσεις, ε, αλλά θέλουμε να ε, ενεργήσουμε και με ευφυΐα. Νομίζω ότι ακούσαμε πολύ καλές εξηγήσει σχετικά με τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Είπατε ότι θα μας υποβάλλετε τα στοιχεία. Θα είναι λοιπόν ε, ένα σημείο ενημερωτικό, θα διανύμουμε τα σχετικά στοιχεία στους Ευρωβουλευτές. Έχουμε κάνει πολλή δουλειά πάνω στον πολιτικό διάλογο για να ξεμπλοκάρουν οι φάκελοι αυτοί. Θα εκτιμούσαμε λοιπόν να λάβουμε περισσότερες πληροφορίες. Σας ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και την ομάδα σας για τις εξηγήσει. Νομίζω ότι κλείνουμε το θέμα αυτό. Καλύψαμε όλες τις παρατηρήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Να αποχαιρετήσουμε τον καλεσμένο μας. So if you all agree... Άψογα.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 Νομίζω ότι έγκαιρα και σύμφωνα με το πρόγραμμά μας έχουμε φτάσει στο σημείο 7 ε, για την αποστολή της αντιπροσωπείας της Επιτροπής, ε, σχετικά με το, της Επιτροπής μας, της Επιτροπής Λιμπής, σχετικά με το δικαστικό σύστημα και τις διαδικασίες ασύλου στην Σουηδία και θα δώσω αμέσως το λόγο στην συνάδελφο Ναταλή Γκρισμπέκ, επικεφαλής αντιπροσωπείας ε, στην Σουηδία και βεβαίως όποιος θέλει μετά μπορεί να πάρει το λόγο μετά την κυρία Γκρισμπέκ. Θα είμαι πάρα πολύ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Πρόκειται για μια αποστολή η οποία έλαβε χώρα πριν από ένα χρόνο περίπου. την οποία έχουμε ήδη εκμεταλλευτεί με την έννοια ότι έχουμε χρησιμοποιήσει ε, την έκβαση αυτών των συζητήσεων και επαφών σε μια σχετική ε, έκθεση. Επομένως ε, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη. Βεβαίως συνήθως όσοι λένε θα είμαι σύντομος μακρηγορούν, αλλά εν πάση περιπτώσει εδώ βλέπω ότι δεν υπάρχουν πλέον πολεμιστές σε αυτή την αίθουσα. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη ε, αποστολή και ευχαριστώ γι' αυτό όλους όσους ε, έλαβαν μέρος σε αυτήν. Ε, είχαμε ενεργή παρουσία, δραστήρια συμμετοχή των συναδέλφων που απέβη ιδιαίτερος χρήσιμη μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα και επομένως είχαμε την δυνατότητα να εμβαθύνουμε ε, στα θέματά μας ε, τα οποία αφορούσαν το δικαστικό σύστημα της Σουηδίας, ε, τις διαδικασίες ε, ασύλου και εστιάσαμε κυρίως, ε, όπως είχαμε συμφωνήσει με τους συναδέλφους, εστιάσαμε λέω κυρίως στο θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Είχαμε την ευκαιρία και την τύχη να συναντήσουμε πολλά πολιτικά πρόσωπα εκπροσώπους των τοπικών αρχών, ε, τοπικούς ερετούς από τους Δήμους ε, της ε, χώρας, καθώς επίσης και πολλούς υπουργούς. Τον Υπουργό Πολιτικής Μετανάστευσης και Ασύλου, κύριο Τομπίας Μπίλστρομ, την Υπουργό Δικαιοσύνης, ε, την ε, Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης ε, και τα λοιπά. Στο υπόμνημα το οποίο σας έχει υποβληθεί έχετε μια πολύ καλή παρουσίαση της αποστολής αυτής. Στη διάρκεια της αποστολής πάντως μπορέσαμε να συζητήσουμε για τα θέματα ασύλου, τον τρόπο κυρίως με τον οποίο ότι οι ξένοι ασυνόδευτοι ανήλικοι ε, ε, ε, λαμβάνονται υπόψη στη Σουηδία, δηλαδή η υποδοχή τους, η παρακολούθησή τους κτλ. Επίσης συζητήσαμε και για το Σουηδικό Δικαστικό Σύστημα καθώς επίσης και την δικαστική συνεργασία. Έχετε την έκθεση, έχετε το υπόμνημα, ενδεχομένως θα μπορούσα να βάλω ε, έτσι εν είδη στιγμάτων κάποια ε, στοιχεία ε, όσον αφορά τη διαδικασία ασύλου στο, στην Σουηδία πρέπει να πω ότι τότε όταν έγινε η αποστολή είχαμε ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα το οποίο δυστυχώς παραμένει στην επικαιρότητα το θέμα της Συρίας και πρέπει να πούμε ότι στην Σουηδία υπήρχε μια μεγάλη εισρωή ε, τον άσυλο από τη Συρία λόγω της ε, σημαντικής ε, συριακής διασποράς στην χώρα αυτή και είδαμε αντίθετα από πολλές άλλες χώρες ότι η Σουηδία είχε ήδη μία οργανωμένη ανταπόκριση για αυτούς τους δυστυχείς Σύριους πρόσφυγες. Όσον αφορά τώρα το ιδιαίτερο ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων που μας απασχόλησε, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε θέλαμε ε, να πάμε στην Σουηδία. Ε, πρέπει να πω ότι είναι εξαιρετικά θετική η εικόνα που αντικατοπτρίζεται όσον αφορά τους ασυνόδευτους ανηλίκους ε, από την Σουηδία, όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των ευάλωτων νέων, όσον αφορά την υποδοχή τους. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Μας έγινε παρουσίαση όλων των οργάνων και των τρόπων ανταπόκρισης που στη Σουηδία δεν βασίζονται ε, όπως τις περισσότερες σε όλες τις υπόλοιπες χώρες ε, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, στην κεντρική κυβέρνηση, αλλά στη Σουηδία βασίζονται στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η κάθε χώρα, συγγνώμη διορθώνω, η κάθε πόλη έχει υποχρέωση να υποδεχτεί συγκεκριμένο προκαθορισμένο αριθμό ασυνόδευτων ανηλίκων. Ε, οι διαδικασίες είναι πολύ συγκεκριμένες, ο τρόπος είναι εξαιρετικά συλλογικός, ε, όλα αυτά μας έκαναν μεγάλη εντύπωση. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει κανένα ε, κατακαιρματισμός, δηλαδή δεν είναι μία υπηρεσία η οποία ασχολείται με την υποδοχή άλλη, με την στέγαση του νέου κτλ. Είναι πολύ συλλογική η δουλειά και επίσης και ένα άλλο στοιχείο το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλες τις χώρες, η ιδιαίτερη αντιμετώπιση αυτής της μεταβατικής περίοδου ανάμεσα ε, στην ενηλικίωση του νέου και την συνέχιση της παρακολούθησης ε, του νέου από τα 18 μέχρι τα 21 του έτη. Ε, δηλαδή άπαξ και ενηλικιωθεί και περάσει τα 18, δεν τον αφήνουν τον νέο μόνο του και ασυνόδευτο. Ε, βεβαίως ε, από ε, δικαστικής απόψεως μας ενδιαφέρει να δούμε πώς μετά τα 18 οργανώνεται η προστασία των νέων αυτών. Εν συμπεράσματι όσον αφορά το σουηδικό σύστημα δικαστικής συνεργασίας μπορώ να πω το εξής. Πρώτα απ' όλα διαπιστώσαμε και όσον αφορά το θέμα αυτό ότι ε, υπάρχουν ε, πολυτομιακές ε, ομάδες οι οποίες εξειδικεύονται κυρίως στα παιδιά, στους ανήλικους. Επίσης ο τρόπος αξιολόγησης, εκτίμησης της ηλικίας είναι πολύ ενδιαφέρον. Στις κάτω χώρες είδαμε παραδείγματα ε, που είναι από τεχνικής άποψης δύσκολα αποδεκτά. Ε, είδαμε επίσης πόσο σημαντικό είναι το θέμα του family tracing και ε, νομίζω ότι είναι και ένα από τα στοιχεία τα οποία ήταν κεντρικά, τα υποβάλαμε στην έκθεση ε, για τους ε, ανήλικους, τους ανήλικους και το δέχτηκαν και όλοι οι συνάδελφοι. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο επίσης και θετικό αυτή η διασύνδεση που ανέφερα και προηγουμένως ανάμεσα στην κεντρική κυβέρνηση, δημοτικές αρχές, συνεργασία ανάμεσα στις αρμόδιες επιτροπές κτλ. Αυτά ήθελα να πω για την αποστολή μας η οποία διήρκε σε δύο μέρες. Ξεκίνησε ξεκίνησε από την Στοκχόλμη ε, και ε, ολοκληρώθηκε στο, στον Δήμο της Σόλνα, στην ευρύτερη περιοχή της Στοκχόλμης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση αυτή που μας κάνατε για την αντιπροσωπεία στη Σουηδία. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Όχι, από ό,τι φαίνεται. Επομένως, να σας ευχαριστήσουμε για μία ακόμα φορά ε, και να προχωρήσουμε ε, με την έκθεση του συναδέλφου Ένση όσον αφορά την επίσκεψη στην Λισαβόνα για το, στο Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών Τοξικομανίας. Αυτή έλαβε χώρα τον Ιούλιο. Έχουμε εδώ τον κύριο Ένση, ο οποίος ήταν και επικεφαλής της αντιπροσωπείας και ο οποίος μπορεί να μας πει δύο λόγια όσον αφορά αυτήν την ε, επίσκεψη της αντιπροσωπείας στη Λισαβόνα. Παρακαλώ κύριε Ένση, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κατάσταση είναι σχεδόν η ίδια. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε πέρσι τον Ιούλιο. Ήταν όμως πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη. Στόχος ε, της αποστολής της ΕΛΥΒΕ ήταν να έχει μια εισβάθος ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις ε, στρατηγικές προτεραιότητες ε, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, του EMCDDA. Εξέτασε το πρόγραμμα εργασίας, την διοίκηση και τον προϋπολογισμό. Είχαμε τη δυνατότητα να συναντηθούμε με τον κύριο Wolfgang Goetz, καθώς και με ε, τον ε, πρόεδρο του Διευθυντικού Συμβουλίου που ε, καθώς επίσης τον, το πρόσωπο που έχει διοριστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκεί πέρα και, άλλους, και άλλα μέλη του Συμβουλίου. Το κέντρο παρακολούθησης δημιουργήθηκε το 1995 και στόχο έχει να παρέχει συμβουλές που να βασίζονται σε επιστημονικά στοιχεία για την διαμόρφωση πολιτικής στον τομέα ε, των ναρκωτικών και της τοξικομανίας. Στόχο έχει επίσης ε, τη συλλογή, ανάλυση και διάδοση πληροφοριών. Το κέντρο παρακολούθηση παρέχει πληροφορίε σχετικά με την κατάσταση των ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά την κατανάλωση και την προσφορά σε συνεργασία με τη Europol. Αναλύει νέε τάσει και παρακολουθεί τις ε, πολιτικές ναρκωτικών των κρατών μελών ε, στο πλαίσιο της ε, ανάπτυξης ευρωπαϊκών πολιτικών. Ωστόσο, το η εντολή του Κέντρου Παρακολούθησης δεν συμπεριλαμβάνει μέτρα που έχουν να κάνουν με τις εθνικές πολιτικές ναρκωτικών των κρατών μελών. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης είχαμε τη δυνατότητα να ακούσουμε παρουσιάσεις εμπειρογνωμόνων του οργανισμού σχετικά με τις βασικές τάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λάβαμε εκτενείς πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο του Κέντρου Παρακολούθησης Εναρκωτικών και Τοξικομανίας όσον αφορά την παρακολούθηση νέων ψυχοτρόπων ουσιών και ιδιαίτερη πηγή ανησυχίας είναι τα λεγόμενα νόμιμα ψυχοτρόπα. Ε, το Κέντρο Παρακολούθησης προσπαθεί να προωθήσει τις βέλτιστες πρακτικές στα κράτη-μέλη Ε, προσπαθεί να, ε, να προσφέρει συμβουλές όσον αφορά τη διαμόρφωση της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συνεργάζεται με μια σειρά διεθνών οργανισμών. Η συνεργασία ανάμεσα στο Κέντρο Παρακολούθησης Τοξικομανίας και ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ φυσικά, αλλά και με τις Επιτροπές Περιβάλλοντος και Προϋπολογισμού. Ήταν, η συνεργασία αυτή είναι επικοδομητική. και η ρύθμιση για τα νέα ψυχοτρόπα μας έδωσε τη δυνατότητα περισσότερων επαφών με το κέντρο αυτό, που παρακολουθεί ακριβώς ε, τις ε, νέες ψυχοτρόπες ουσίες που αποτελούν κεντρικό κομμάτι της νέα νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό λυπάμαι που ο προϋπολογισμός του κέντρου έχει μειωθεί κατά 5% για το 2014. Αν σκεφτούμε τη σημασία της εξαιρετικής δουλειάς και εμπειρογνωμοσύνης που παρέχει πάνω στην διακίνηση και ε, κατάχρηση ναρκωτικών. Τα φαινόμενα αυτά απειλούν την υγεία των πολιτών μας και ιδιαίτερα των νέων. Έτσι απειλούν την σταθερότητα των κοινωνιών μας. Η ποιότητα της δουλειάς του κέντρου μας δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη για περισσότερη ορατότητα της δουλειάς που κάνει το Κέντρο Παρακολούθησης ε, Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Θα πρέπει να επιδιώξουμε μια πιο στενή συνεργασία ανάμεσα στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ του Κοινοβουλίου και το Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας. Αυτά. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστώ. Υπάρχουν σχόλια μετά την παρουσίαση για την επίσκεψή μας στη Λισαβόνα στην ε, Οργανισμό για τα Ναρκωτικά. Ευχαριστούμε κύριε Ένσιου για την παρουσίαση και την επίσκεψη. Και το τελευταίο σημείο μας πριν την συνεδρίαση των συντονιστών που βλέπετε στις 11.30 θα έχουμε μια παρουσίαση από τον κύριο Τερί Σούλμπρεκ που εκπροσωπεί την εταιρεία Lloyd Belgium και ξεπώνησε μια έκθεση για τη χρηματοδότηση που δίνει η Ένωση σε μη κυβερνητικέ οργανώσει για τι εσωτερικέ υποθέσει, την ασφάλεια και τη μετανάστευση. Αυτό θα προκαλέσει και κάποια συζήτηση. Κύριε Φανσούμπρεκ, ε, καλώς ήρθατε. Παρακαλώ ε, να ακούσουμε την παρουσίασή σας ε, για το θέμα αυτό. Σύντομη εισαγωγή. Να σας θυμίσω τους στόχους της έκθεσης, ε, διαφάνεια, για το πώς λειτουργεί η χρηματοδότηση μη κυβερνητικών οργανώσεων για τις εσωτερικές υποθέσεις, την ασφάλεια και την μετανάστευση. Τέσσερις μελέτες, ε, γενικές αρχές χρηματοδότησης ε, της Ένωσης, ποσοστοποίηση, ποσοτικοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων που χρηματοδοτούνται κεντρικά, το διοικητικό βάρος που αντιμετωπίζουν μη κυβερνητικές οργανώσεις για να εφαρμόσουν ε, τις υποχρεώσεις που προκύπτουν με τη χρηματοδότηση και τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ληφθεί από την Επιτροπή για να υπάρξει περισσότερη αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και διαφάνεια. Μελετήσαμε όλες τις σχετικές μελέτες, συζητήσαμε με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς για την ποσοτικοποίηση, είδαμε τα στοιχεία για τη χρηματοδότηση που υπάρχουν στο σύστημα για την ε, χρηματοδοτική διαφάνεια και στο κοινό μητρό για τη διαφάνεια. Και βασιστήκαμε και σε στοιχεία που μας έδωσε για, τα λογιστική, για τη λογιστική πλευρά του θέματος, η Γενική Διεύθυνση για τον Προϋπολογισμό επίσης. Μελετήσαμε και 10 περιπτώσεις μη κυβερνητικών οργανώσεων, Κάριτας, Διεθνής Διαφάνεια, ε, το Ίδρυμα για την ε, Μελέτη, για την ισότητα των φύλων και ε, ο Οργανισμός για τη Βοήθεια στα Θύματα της Δημοκρατίας. Πρώτο λοιπόν, οι αρχές της χρηματοδότησης της Ένωσης για μη κυβερνητικές οργανώσεις. Επειδή δεν υπάρχει νομικός ε, ορισμός ε, επίπεδο ένωσης ε, της μη κυβερνητικής οργανώσεως, το τι είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση δεν έχουμε αρκετά εύκολα προσβάσιμη πληροφόρηση. Δεν είναι βεβαίως αμεληταίο το ποσοστό της χρηματοδότησης που παίρνουν μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά δεν υπάρχει νομική υποχρέωση να το αναφέρουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσει αντιμετωπίζονται τον ίδιο τρόπο με οποιονδήποτε άλλο λαμβάνει χρηματοδότηση. Ποιο είναι το θέμα. Το FTS δεν έχει πληροφόρηση για τις μη κυβερνητικέ οργανώσει χωριστά και στο κοινό μητρό για τη διαφάνεια είναι εθελοντική η συμμετοχή, άρα είναι ανεπαρκές για βάση. Το σύστημα ABAC της Ένωσης, το εσωτερικό σύστημα χρηματοδοτικής πληροφόρησης μπορεί να μας ενημερώσει για στοιχεία για, τις, για τους μη οργανισμούς και για τις μη κερδικές οργανώσεις, αλλά τώρα άρχισε να λειτουργεί το 2013, άρα δεν έχουμε στοιχεία, συστάσεις. Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε έναν διοργανικό διάλογο για να καταλήξουμε σε έναν ενωσιακό ορισμό του τι σημαίνει μη κυβερνητική οργανώση, όχι τόσο πολύ για νομικούς, αλλά για λόγους ε, συλλογής στοιχείων. Αν είχαμε έναν ε, ευρέως ε, αποδεκτό ορισμό, θα μας βοηθούσε να ελέγξουμε τη χρηματοδότηση, άρα θα αυξήσει τη διαφάνεια. Να συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειες, να βελτιωθεί το FTS και το JTR, δηλαδή το κοινό μητρό διαφάνειας θα μπορούσαμε έτσι να λάβουμε περισσότερα στοιχεία από το σύστημα της Κομισιόν ΑΜΠΑΚ. Δεύτερο σημείο. Ποια είναι τα ποσά της βοήθειας που λαμβάνουν μη κυβερνητικέ οργανώσεις, από ό,τι βλέπουμε, από τους πόρους ε, που είναι αντικείμενο κεντρικής διατήρησης, το 2010 είχαμε 12 ε, εκατομμύρια, το 2011 11,9 και το 2012 30 εκατομμύρια. Χρειάστηκε να δω ε, σελίδα σελίδα όλη τη χρηματοδότηση που υπάρχει στο FTS και ούτως ή άλλως 90% της χρηματοδότησης δίνεται με κοινό σύστημα διαχείρισης. Η χρηματοδότηση αφορά και τις λειτουργικές δαπάνες, διοικητικές δηλαδή. Η Γενική Διεύθυνση Home εφαρμόζει παντού το όριο του 7% αποζημίωσης για διοικητικό κόστος. Αν το συγκρίνουμε με άλλους θεσμικούς δωρητές στον τομέα των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η Ελβετία για παράδειγμα, βλέπουμε ότι και αυτή δέχονται ποσοστά χρηματοδότηση των διοικητικών δαπανών 5-18%. Αν δούμε συνολικά το διοικητικό κόστος ε, που συμπεριλαμβάνει και την ενημέρωση και την προσπάθεια συλλογής πόρων βλέπουμε ότι είναι στο 9-15% σε σχέση με αυτό. Όπως ήδη είπα, θα ήταν καλύτερα να έχουμε καλύτερη σηματοδότηση των οργανώσεων αυτών και το ανώτατο όριο του 7% για τις επιστροφές νομίζουμε ότι είναι περίπου κατάλληλο για τις ανάγκες τους είναι λίγο χαμηλότερο από το πραγματικό τους κόστος έτσι τους ε, ενθαρρύνουμε να έχουν πιο αποτελεσματική διαχείριση. Τι διοικητικό τώρα βάρος σημαίνει αυτό για τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. 9 από τις 10 περιπτώσεις που εξετάσαμε αναλυτικά μας είπαν επανειλημμένα ότι το διοικητικό βάρος είναι σημαντικό εμπόδιο για να ε, κάνουν αίτηση και να λάβουν ενωσιακή χρηματοδότηση. Όσο μεγαλύτερο είναι το ε, διοικητικό βάρος, τόσο μεγαλύτερο είναι και το ποσοστό των πόρων που τελικά δεν χρησιμοποιείται για τον πραγματικό σκοπό των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Βεβαίω, ο νέο ε, δημοσιονομικό κανονισμό έχει βελτιώσει την κατάσταση, αλλά παραμένουν κάποια προβλήματα θα παρακαλούσαμε την ε, Γενική Διεύθυνση Home να εντείνει το διάλογο με τις ΜΚΟ για να καταλάβει τι σημαίνουν οι διαδικασίες της για τις ΜΚΟ και να τους δώσει περισσότερη βοήθεια απλοποιώντας τις διαδικασίες. Επίσης να δουν το ενδεχόμενο τα συστήματα διαχείρισης ε, των διαφόρων επιδοτήσεων των διαφόρων γενικών διευθύνσεων να είναι πιο συντονισμένα, ευθυγραμμισμένα. Γιατί πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, ζητούν από διάφορες γενικές διευθύνσεις χρηματοδοτήσεις και άρα πρέπει να αντιμετωπίσουν διάφορα συστήματα. Με βάση τα προγράμματα τώρα για το 2014 και 2020 έχουμε τη σύσταση να υπάρχει πολιετής χρηματοδότηση για τις ΜΚΟ, γιατί έτσι έχουν περισσότερη χρηματοδοτική ασφάλεια να υπάρχουν κοινοί κανόνες για τα προγράμματα χρηματοδότησης. Αυτό δεν διευκολύνει διαδικαστικά και να υπάρχουν πιο ευέλικτοι μηχανισμοί για να αντιμετωπιστούν επίγουσες απρόβλεπτες καταστάσεις. Τελευταίο θέμα, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της χρηματοδότησης των ΜΚΟ. Είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί κανόνες και διαδικασίες που ήδη υπάρχουν για να διασφαλιστεί, να διασφαλιστεί η ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα Ωστόσο, οι μελέτες που έγιναν και όπως ε, ανέφεραν και διάφοροι φορείς με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή, υπάρχουν αδυναμίες. Δεν δίδεται επαρκής ε, πληροφόρηση εκ των υστέρων για το τι έγινε με την αίτησή τους. Επίσης, θα μπορούσε η συγχρηματοδότηση να γίνεται σε είδος για παράδειγμα, να κοστολογηθεί η συμμετοχή ε, εθελοντών. Αυτό θα οδηγούσε σε μικρότερες ε, επιδοτήσεις. Δεν έχουν επίσης επαρκή εξοπλισμού και γνώση οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να αποτιμήσουν την εργασία τους και την απόδοσή της και τέλος, αλλά όχι δεν αξιοποιείται αρκετά από τις υπηρεσίες δεν αξιοποιούνται οι εκθέσεις που κάνουν οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις για το πώς πήγαν τα προγράμματά τους. Αυτό θα έπρεπε να δίδεται ως δυνατότητα σε όλες τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις να κάνουν τέτοιες εκθέσεις γιατί αυτό θα μας, θα μας ωφελούσε όλους. Αυτή είναι η εισαγωγή μου. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαν για την ε, παρουσίαση που μας κάνατε όσον αφορά τις ε, μη κυβερνητικούς ε, οργανισμούς. είχαμε προβλέψει και συζήτηση, οπότε έχουμε χρόνο. Κύριε Πίρκελ, παρακαλώ. Πρόεδρε. Χαίρομαι πάρα πολύ που εκπονήθηκε η μελέτη αυτή, διότι είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν οι πόροι που διατίθενται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιούνται με το βέλτιστο τρόπο. Υπάρχει λοιπόν μεγάλο ενδιαφέρον σχετικά με το πώς, πόσα κονδύλια πηγαίνουν ε, σε, για διοικητικές δαπάνες και πόσο μεγάλο μέρος των ε, κονδυλίων δαπανάται ε, σε προγράμματα. Και από πλευράς της Κομισιόν θα υπάρξει βελτίωση, δηλαδή θα μειωθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια και θα έχουμε περισσότερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Αυτή ήταν η στόχη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την μελέτη αυτή. Είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε επανειλημμένα και είναι πολύ ενδιαφέρον που έχουμε μπροστά μας τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής. Αναφέρονται κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα μη κυβερνητικών οργανώσεων, διότι δεν υπάρχει φυσικά η δυνατότητα να αναφερθούν όλες, αλλά έγινε ανάλυση της κατάστασής τους και έχουν εξαχθεί ε, συμπεράσματα, τα οποία απευθύνονται και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε εμά ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σα ευχαριστώ λοιπόν πολύ. Δύο ερωτήσει έχω. Η πρώτη ερώτηση είναι. Βλέπουμε ότι οι πόροι που αναφέρονται έχουν να κάνουν Είδαμε ότι οι πόροι προ τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις ε, έχουν ε, αυξηθεί από 12 εκατομμύρια ευρώ σε 30,1 εκατομμύρια ευρώ μέσα σε δύο χρόνια. Σχεδόν ε, έχουν τριπλασιαστεί οι πόροι. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις έχουν λάβει τριπλάσιου πόρου μέσα σε δύο χρόνια. Η δεύτερη ερώτηση είναι διαφορετική. Είπαμε ότι μόνο συγκεκριμένε μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, μπορούν να εξεταστούν. Εξετάσατε μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, που ενεργούν σε εθνικό επίπεδο και που λαμβάνουν και σε εθνικό επίπεδο πόρου. Είναι γεγονός ότι το 20% των πόρων διατίθεται με αυτό το direct management, επειδή ακριβώς τα προγράμματα αυτά οργανώνονται σε κεντρικό επίπεδο. Αυτή είναι η προϋπόθεση. Αλλά το 80% διοχετεύεται μέσω εθνικών προγραμμάτων που δεν ε, καλύπτονται από τη μελέτη. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι, προσπαθήσατε να λάβετε πληροφορίες και από τους υπεύθυνους σε εθνικό επίπεδο αυτούς που είναι υπεύθυνου για τα εθνικά προγράμματα. Υπήρξαν προβλήματα κατά τη συλλογή τέτοιων πληροφοριών και γνωρίζετε εάν υπάρχει κάποια επισκόπηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με το τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχει ο ίδιος βαθμός διαφάνειας, υπάρχουν τα ίδια ανώτατα όρια κονδυλίων για τα προγράμματα έχουμε εμείς ακριβώς αυτή την οροφή του 10% το ανώτατο όριο. Τι ισχύει λοιπόν για το 80% των πόρων που διατίθενται σε εθνικό επίπεδο. Δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Έχετε εσείς τέτοιες πληροφορίες. Σε εθνικό επίπεδο είναι η ίδια η κατάσταση ή διαφορετική. Και μπορείτε να συλλέξετε πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα που πραγματοποιούνται σε εθνικό επίπεδο. Σα ευχαριστώ πολύ. κυρία Κιγιόμ. Και εσείς έχετε τον λόγο κυρία Κιγιόμ. ναι, ούτως ή άλλως δεν είμαστε και πολλοί. Δεν θα επανέλθω επί της ουσίας γιατί ζητώ συγγνώμη αλλά δεν διάβασα ε, τι λεπτομέρειές της την έκθεση αυτή την οποία προτίθεμαι να διαβάσω. Επομένως δεν θα μπορούσα να κάνω ε, επί της ουσίας παρατηρήσεις. Επί του τύπου όμως, της μορφής. Μιλήσαμε προηγουμένως με τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα πρώτα στάδια της ε, υλοποίησης εθνικών προγραμμάτων όσον αφορά τα ταμεία τα οποία σχετίζονται ε, με θέματα δικαστικά και εσωτερικών ε, υποθέσεων και επομένως ε, βλέπουμε, ε, έχοντας συζητήσει με τα κράτη-μέλη, τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη σε σχέση με την προώθηση χρηματοδότησης προς τις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Αλλά να σας πω ότι εμείς προσπαθήσαμε να τροποποιήσουμε τους κανονισμούς, τους χρηματοδοτικούς κανονισμούς. Ψηφίσαμε πριν από λίγο καιρό. Παρ' αυτά έχω την εντύπωση ότι υπάρχει μία διάσταση με αυτά που μας προτείνετε εσείς τώρα γιατί διαφορετικοί κανόνες, διοικητικά ε, ε, δυσκινησίες γραφειοκρατικές, προθεσμίες, όλα αυτά τα συζητήσαμε και πριν. Φαντάζομαι ότι χρήσιμο θα ήταν να έχουμε βέβαια αυτά τα ε, στοιχεία ανάλυσης, αλλά κυρίως κάποιες συστάσεις από τη δική σας πλευρά όσον αφορά τον την τροποποίηση πούμε, του χρηματοδοτικού κανονισμού ή μιας διαφορετικής χρηματοδοτικής αντιμετώπισης ε, να κάνετε κάποιες ε, συστάσεις και να τις αναλύσετε. Εδώ ε, μας, δώσ, μας δείξετε τις διαφάνειες αυτές, οπότε φαντάζομαι ότι μελετώντας ε, θα βρω κάποια τέτοια παραδείγματα. Αλλά κυρίως αφού έχετε ολοκληρώσει και εσείς την εργασία σας βλέπετε να υπάρχει ευθεία αντιστοίχηση με τη δική μας εργασία όσον αφορά τους κανονισμούς. Σας ξαναδώσω το λόγο κύριε Βαν Σούρμπροκ για να απαντήσετε ένα σχόλιο πρώτο όσον αφορά την τελευταία ερώτηση η οποία σχετίζεται με, την, ε, ε, με τη χρονική στιγμή της ε, ε, μελέτης. Ε, πρέπει να σας πω ότι η ανάθεση έγινε το τέλος του προηγούμενου χρόνου, επομένως ε, εργαστήκαμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα πώς αυτό το χρονοδιάγραμμα καλύπτει η έντιστοιχή με το δικό σας χρονοδιάγραμμα, δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσα να ελέγξω. Σχετικά με τα σχόλια που έκανε ο κύριος Πίρκελ για την αύξηση των ποσών ε, και όσον αφορά την κεντρική ε, άμεση χρηματοδότηση, ε, νομίζω ότι ο Λιονέλ μπορεί να απαντήσει από αυτού. Είδαμε να αυξάνονται όντως τα ποσά δεν υπάρχει ιδιαίτερη εξήγηση. Αυτό σχετίζεται κυρίως με τα διάφορα προγράμματα τα οποία αξιολογήσαμε από την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς επίσης ε, και ε, με την χρηματοδότηση την οποία διαπιστώσαμε. Και βεβαίω ε, αυτή η χρηματοδότηση δεν αφορά μονάχα μη κυβερνητικέ οργανώσει, έχει και άλλου δικαιούχου που του καθορίζουν τα κράτη-μέλη. Είναι πιθανό στην τελευταία προγραμματική περίοδο τα ποσά τα οποία ανατέθηκαν ε, στις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, διατέθηκαν μάλλον μη κυβερνητικέ οργανώσεις, ήταν πιο μεγάλα από αυτά που δόθηκαν σε άλλους φορείς. Και για να επανέλθω και στην άλλη ερώτηση όσον αφορά αυτήν την, ε, αυτά τα ποσοστά του 80-90% που διαχειρίζονται τα κράτη-μέλη άμεσα, ναι, είναι γεγονός ότι ε, η διαχείριση γίνεται περισσότερο ε, σε ευρωπαϊκό ε, επίπεδο, αλλά ξέρετε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει πλέον αυτό το σύστημα ε, διαφάνειας μέσω του οποίου δίνονται τα χρήματα, τα κονδύλια και στις μη κυβερνητικές οργανώσεις και στους υπόλοιπους δικαιούχους μέσω των Υπουργείων. Ε, αυτό σημαίνει ότι τα Υπουργεία και οι ενδιάμεση φορείς ε, πρέπει να έχουν την υποχρέωση να δημοσιοποιούν όλα τα στοιχεία, αλλά δεν υπάρχει ενιαίος κατάλογος ε, και εν πάση περιπτώσει και οι φυστάμενοι κατάλογοι δεν είναι πάντα απολύτως επικαιροποιημένοι. And, uh, yeah, uh, uh, Και τέλος, παράδειγμα σύστασης το οποίο δίνουμε όσον αφορά την ποσοστοποίηση της χρηματοδότησης των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα ορισμός ε, όσον αφορά, σε ενωσιακό επίπεδο όσον αφορά ε, την, ε, το σαφές reporting, τη σαφή υποβολή εκθέσεων. Θα πρέπει πρώτα να καθοριστούν, να υπάρξει δηλαδή ορισμός των μη κυβερνητικών οργανώσεων έτσι ώστε να υπάρχει και η δυνατότητα ποσοστοποίησης όλων αυτών των στοιχείων. Επομένως και με τον τρόπο αυτό και εάν όλες οι πληροφορίες ήταν ε, διαθέσιμες στο Μητρό Διαφάνειας, βεβαίως θα βελτίωνε περισσότερο την διαφάνεια όσον αφορά τη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ωραία. Ε, στα πλαίσια του ετήσιου προγράμματος ε, ε, της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών είχαμε καταγράψει, είχαμε εγγράψει μάλλον σε αυτό το πρόγραμμά μας και την μελέτη για την έκθεση αυτή, οπότε πολύ ωραία. Τώρα έχουμε όμως την των, τη συνεδρίαση των συντονιστών, αλλά σε 15 λεπτά από τώρα στις 11.30. Είναι σημαντική, έκθεση, σημαντική η συνεδρία των συντονιστών γιατί θα συζητήσουμε για τις εκθέσεις, ποιος θα κάνει τι κτλ. Ε, πολύ ωραία. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα λάβει χώρα στις Βρυξέλλες την 31η Μαρτίου και την 1η Απριλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για την παρουσία σας και τη συνεργασία σας και σας χαιρετώ.